Κύριε Μάνκα, είσαστε συνεισηγητής. Ο άλλος συνεισηγητής έρχεται. Ε, πρέπει να αρχίσουμε, γιατί έχουμε 60 λεπτά στη διάθεσή μας για τη συζήτηση αυτή. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε και σύντομοι στις παρεμβάσεις μας. Οπότε, αν συμφωνείτε κι εσείς, κυρίσω την έναρξη της συνεδρίασης αυτής. Συγγνώμη ζητάει ο Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη, ο οποίος έχει άλλες ανελημμένες υποχρεώσεις και ο οποίος θα έρθει κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ημερήσια διάταξη. Συμφωνείτε, υπάρχουν παρατηρήσεις. Εγώ δεν έχω ανακοινώσεις, οπότε θα δώσω το λόγο για 5 λεπτά σε έκαστο εκ των δύο συνεισηγητών. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Μάνκα παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και είναι παράδοξο ότι ναι μεν είμαι συγητής αλλά δεν έχω διαρμηνία στην ίδια μου τη γλώσσα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδες συζήτητες οι, οποίες, ε, οι οποίοι παραβρέθηκαν στις συνεδριάσεις μας και μας βοήθησαν να δημιουργήσουμε μια ατμόσφαιρα κατά την οποία όλοι αισθάνονταν ότι μετρήσε η κάθε άποψη. Και εμείς ως εισηγητές μαζί με τους ε, συμβούλους μας εξετάζουμε κάθε γνώμη και εξετάζουμε τους τρόπους ε, εξεύρεσης συνένεση σε κάποιες ε, ομάδες των οποίων οι εκπρόσωποι ήθελαν να καταψηφίσουν την έκθεση καθεαυτή, πλέον να ζητούν κοινέ λύσεις μαζί μας. Αυτό είναι πολύ θετικό. Να συνεχίσουμε λοιπόν, ελπίζω, αύριο στην συνάντηση των σκιωδών εισηγητών και νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο για να βρούμε καλές λύσεις. και θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο για να συνεχίσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και να ευχαριστήσω και εγώ του συναδέλφου. Να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Μάνκα, τον συνεισηγητή μου, για την ε, πολύ καλή συνεργασία και την ε, πολύ καρποφόρο εργασία των τελευταίων εβδομάδων εν ώψη και της προετοιμασίας των συμβιβασμών. Τα συζητάμε λοιπόν αυτά ήδη με τους κοιόδες μας. Και όπως θα θυμάστε, το σχέδιο της έκθεσης το οποίο παρουσιάσαμε, ενώ είναι ρεαλιστικό, λαμβάνει υπόψη είναι αφενός τις διαφορετικές απόψεις που επικρατούν για το θέμα αυτό και αφετέρου το τρέχον πολιτικό σκηνικό και τις προτεραιότητες που χαρακτηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν η πρόταση των συνεισηγητών για τη μεταρρύθμιση του ESM βασίζεται σε μία διπλή ε, προσέγγιση. Μία βραχυπρόθεσμη πρώτος και σε μακροπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο επίπεδο να ξεκαθαρίσουμε ποιες είναι οι προτεραιότητές μας. Λάβαμε 237 ε, τροπολογίες στην αρχική μας πρόταση. Καλύπτουν πολλά διαφορετικά πολιτικά ζητήματα και θέματα τα οποία είναι σε διαφορετικό βαθμό αμφιλεγόμενα, αλλά ουσιαστικά επικεντρωνόμαστε σε τέσσερα βασικά στοιχεία, τα οποία θεωρώ ότι θα αποτελέσουν και την καλή βάση για την εξεύρεση συμβιβαστικών λύσεων μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Έχουμε λοιπόν ήδη μία, είχαμε μια πρώτη ε, επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων. Μια δεύτερη προγραμματίζεται για αύριο θα ήθελα να τονίσω σε ό,τι αφορά τον όγκο των τροπολογιών το εξή. Η πρώτη ομάδα τροπολογιών έχει να κάνει με την ανάγκη να εξασφαλίσουμε και βραχυπρόθεσμα ακόμα συγκεκριμένες φιλόδοξες δράσεις για να ενισχυθούν τα θέματα νομιμότητας, δημοκρατικής νομιμότητας και λογοδοσίας στο Κοινοβούλιο. Κάποιες τροπολογίες λοιπόν θέλουν ερωτήσεις, θέλουν να ζητήσουν, να ζητούν ακροάσεις, δικαιώματα διορισμού και δικαιώματα ελέγχου προπολογισμού σε ό,τι αφορά τη διαδικασία χορηγή απαλλαγή. Οι συνεισηγητέ είμαστε πολύ υπέρ τη ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου, ενώ παράλληλα θέλουμε να σεβαστούμε και την διακυβερνητική φύση του σώματος αυτού και θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε έβρεση ευρείας ε, συνένεση στο θέμα αυτό. Επίσης, θα χρησιμοποιήσουμε και το προτινόμενο μνημόνιο συμφωνίας ε, ως εργαλείο για να βελτιώσουμε το ρόλο του Κοινοβουλίου. Επίσης, υπάρχει ευρεία συμφωνία και υποστηρίξη για την ιδέα της μελλοντική ε, μεταρρύθμισης του πλαισίου αυτού στο νομικό πλαίσιο. Είναι σαφή η άποψη του Κοινοβουλίου και θα θέλαμε να συνεχιστεί αυτή η υποστήριξη. Μία δεύτερη ομάδα τροπολογιών τώρα έχει να κάνει με το όνομα του μελλοντικού σώματος της υπηρεσίας αυτής. Και εδώ ξέρετε ότι έχουμε παρουσιάσει μία πρόταση και φαίνεται ότι δεν υπάρχει πολιτική υποστήριξη ενία για το θέμα αυτό παρά το γεγονός ότι υπάρχει ευρεία συμφωνία με την ιδέα ότι το όνομα της υπηρεσίας αυτής δεν θα πρέπει να είναι Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι θα υπήρχε, όπως και να το κάνουμε, μια άλλη επικάλυψη με τις ε, ε, αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η απόψη των εισηγητών, των σκιωδών. Κατά πάσα πιθανότητα θα παραμείνει κρεμές το θέμα αυτό. Τρίτη ομάδα τροπολογιών σε ό,τι αφορά την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωζώνης γιατί θέλουμε μια ισορροπία μεταξύ αλληλεγγύη και υπευθυνότητα και θα θυμάστε. Η συνθήκη ESM ήδη πρότεινε μια σύνδεση με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Μακροοικονομικής ε, Εποπτείας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά και το πακέτο, το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, έχοντας υπόψη και τις, ε, τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου, πιστεύω ότι θα πρέπει να περιοριστούμε στο τρέχον νομικό πλαίσιο και να επεξεργαστούμε τη βάση αυτή. Η τελευταία ομάδα τροπολογιών έχει να κάνει με τα εθνικά κοινοβούλια και το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων. Και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προφανώ. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτή την προσέγγιση σε δύο βήματα ότι ενώ πρόκειται για διακυβερνητικό σώμα και ο ρόλος του Κοινοβουλίου των Εθνικών προφανώς θα πρέπει να διατηρηθεί και να βελτιωθεί αν λάβουμε υπόψη μια πιο μακροπρόθεσμη α, προοπτική όπου θα υπάρξει μια ένταξη ενδεχομένω στο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο, ο ρόλος του Κοινοβουλίου λοιπόν στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να βελτιωθεί, το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. αλλά και βράχει πρόθεσμα. Πιστεύουμε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωση ό,τι αφορά το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτά λοιπόν είναι τα ζητήματα τα οποία επεξεργαζόμαστε στις τροπολογίε μας. Τα συνεργαστούμε στενά για να πετύχουμε ένα συμβιβασμό και πραγματικά πιστεύω ότι αυτό είναι εφικτό. Και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρο, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Συνεισηγητή για τι διευκρινήσει αυτέ. Πολύ ενθαρρυντικά τα όσα μα λέτε για να πετύχουμε ένα συμβιβασμό και έγκριση στην ε, Ολομέλεια τη έκθεση πρωτοβουλία αυτή. Και τώρα να βάζω το λόγο στου σκιώδει εισηγητέ από την Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού και την ομάδα του ΕΛΚ. Ο κύριος Μούρας αν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. ευχαριστώ πολύ τους δύο συνεισηγητές, τους συναδέρφους μας, τον κύριο Μάνκα και τον κύριο Σίλβα Περέιρα, για το σχέδιο αυτό έκθεσης που πρέπει να πω ότι αποτελεί μια πάρα πολύ καλή βάση προς συζήτηση. Χρειάζονται κάποιες διορθώσεις, κάποιες τροποποίησεις πιστεύω, αλλά γενικά μιλώντας έχω την αίσθηση ότι οι συναντήσεις με τους κοιόδες εισηγητές είναι ιδιαίτερα επικοδομητικές και θα καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν εμείς πρέπει να περάσουμε ένα σαφές μήνυμα. Και γι' αυτό και θα ήθελα η έκθεση να παραμείνει σύντομη και συνοπτική. Και το λέω αυτό και εκ μέρους του ΕΛΚ και γι' αυτό και περιόρισα τις τροπολογίες μας και στην Επιτροπή Προπολογισμών για να διατηρηθεί ο σύντομος χαρακτήρας της έκθεσης αυτής. Τροπολογίες θα έχω για πράγματα που πιστεύω ότι πρέπει να ενισχύσουμε και λείπουν. Πρώτα απ' όλα, οι συνεισηγητές είπαν ότι πρέπει να συμμορφωνόμαστε με τους κανόνες και τις υποχρεώσεις μας. Εδώ υπογραμμίζω τη σημασία που έχουν οι δημοσιονομικοί κανόνες. Πρέπει να υπάρχει δημοσιονομική προστασία ώστε να μην είμαστε ευάλωτοι σε κακές στιγμές. Όλοι γνωρίζουμε ότι το έλλειμμα και το πλεόνασμα είναι πράγματα τα οποία επηρεάζονται σε καλές και σε κακές στιγμές. Επίσης, θα ήθελα να πιέσω και για διορθωτικές αλλαγές, που σημαίνει άνοιγμα της οικονομίας, μείωση του κόστους και θυσίες που πρέπει να γίνουν σε περίοδους κρίσης. Πιστεύω ότι ό,τι κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις ευθύνε και τις αρμοδιότητες σε εθνικό επίπεδο. Αυτά που κάνουμε εμεί είναι πολύ σημαντικά. Σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν ε, κάποια δίκτυα προστασίας, δημοσιονομικές ε, πολιτικές που πρέπει να είναι σωστά και να χρησιμοποιούνται καλά με τα σωστά εργαλεία για να πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Επίσης, χρηματοδότηση για ε, περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Και αυτό πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας και στα πλαίσια του ESM. Πρέπει να συμπεριληφθεί στις συνθήκες το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, πιστεύω. Και έχω και τροπολογία που λέει ότι οι χώρες που δεν είναι στην ΟΝΕ να μπορούν να συμμετέχουν και μετά το Brexit μόνο η Δανία θα έχει opt-out από το ευρώ. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να διευκολυνθεί η σύγκληση αυτή. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να σας πω ότι είναι καλό που το ετοιμάζουμε το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Χωρίς αυτό είναι πιο αδύναμο το κοινό μας νόμισμα και ανεπαρκές. Σίγουρα υπάρχουν ε, κάποιες αδυναμίες ακόμα, αλλά γι' αυτό πρέπει να κάνουμε καλά αυτή τη δουλειά. Ξέρουμε σήμερα τι δεν κάναμε καλά πριν από 20 χρόνια και γι' αυτό τώρα πρέπει να το κάνουμε σωστά και να μην είναι μόνο μια πολιτική απόφαση. Με την έκθεση των συναδέρφων και με τις τροπολογίες πιστεύω πραγματικά, Πρόεδρε, ότι θα καταλήξουμε σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ κύριε Μουρεσάν. Τώρα το λόγο έχει ο Τόμ Βαντεκάντελλαρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ του συνεισηγητές για την έκθεση αυτή και τον συνάδελφο Μουρεσάν. Ε, και εγώ έχω δουλέψει μαζί του στο ΕΛΚ. Πιστεύω και εγώ ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα καλό συμβασμό, αλλά πρέπει και να βιαστούμε χρόνος, γιατί πιέζει ο χρόνο. Μου άρεσε η αρχική έκθεση. Πιστεύω ότι πρέπει βέβαια να υπογραμμίσουμε κάποια σημεία και να γίνουν διαπραγματεύσεις τα εξή. Πρώτον, όσον αφορά τις προϋποθέσεις, νομίζω ότι είναι γνωστό ότι η ομάδα μας, πράγματι όπως είπε και ο συνάδελφος Μούρισαν, εδώ πέρα πρόκειται για βοήθεια σε περίπτωση κρίσης. Οπότε πρώτα απ' όλα αυτό που θέλουμε είναι οι χώρες μέλη πρώτα απ' όλα να βάλουν τάξη στα του οίκου τους πριν περάσουμε στο ταμείο. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει όντω να βάλουμε τις προϋποθέσεις και να είναι πιο αυστηρές. Εξάντε προϋποθέσεις να υπάρχουν πρώτα απ' όλα ε, καλή ε, οικονομική κατάσταση, αλλά να λάβουμε υπόψη μας και κάποιες ex post προϋποθέσεις. Ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ας πούμε, σε περίπτωση κρίσης. Έπειτα, ο κύριο Σίλβα Παρέρα αναφέρθηκε στην δημοκρατική νομιμότητα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά την εποπτεία από πλευρά των Εθνικών Κοινοβουλίων. Πολύ χαιρόμαστε που τα Εθνικά Κοινοβούλια αναφέρονται στην έκθεση αυτή. Για μας είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι θέλουμε την ε, δημοκρατική αυτή εποπτεία από τα Εθνικά Κοινοβούλια, δεν θέλουμε να τη θάψουμε. Έπειτα, οι χώρε μέλη είναι ε, εκείνες που θα προσφέρουν στο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Τομείο και το, κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρέπει να υπάρχει δικαίωμα να γνωρίζουμε τι ακριβώς κάνει το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Πρέπει να μπορεί να υπάρχει διάλογος δηλαδή μαζί τους δημοκρατική νομιμότητα λοιπόν και ο ρόλος των ηθικών κοινοβουλίων. Αυτό ήταν το δεύτερο σημείο. Τρίτο, η ονομασία. Μπορούμε να στηρίξουμε τους φιλελεύθερους συναδέρφους να μείνουμε στο μηχανισμό σταθεροποίησης και όχι στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι για Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. δεν πρέπει να υπάρχει πολύ έντονα αυτή η νομισματική πτυχή. Οπότε αυτό ήταν το όνομα, το τρίτο σημείο. Και το τελευταίο μου σημείο έχει να κάνει με άλλες συζητήσεις. Το έχουμε πει ότι πρέπει να μείνουμε όσο γίνεται πιο κοντά στο αρχικό κείμενο. Ε, ναι, με διάφορες τροπολογίες μπαίνουν και άλλα θέματα, προστίθενται κτλ. Αλλά ένα βασικό σημείο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να παραμείνουμε όσο γίνεται πιο κοντά στο αρχικό κείμενο. για τις δημοσιονομικές ικανότητες, για τους υπουργούς οικονομικών, για τον προπολογισμό της ε, ε, Ευρωζώνης. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία μας προβληματίζουν, αλλά δεν έχουν θέση εδώ και δεν θα μπορέσουμε, αν πρέπει να συζητήσουμε και για όλα αυτά, να τηρήσουμε και το χρονοδιάγραμμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπεν Κόλμελ κανονικά έχει σειρά, δεν τον βλέπω όμως. Ο συνάδελφός του έχει λόγο. Από πλευράς ECR, ο Ραλφ Πάκετ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συγγητές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να συμπεριλάβουμε των Πεκών Μηχανισμού Σταθερότητα στο νομικό πλαίσιο Ευρωπαϊκή Ένωση και να αλλάξει η ονομασία σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο θα αναλάβει ήδη τι λειτουργίε του μηχανισμού σταθερότητα, αλλά έχει νέα διοίκηση σε κεντρικό επίπεδο. Δεν συμφωνώ με αυτή την προσέγγιση, γι' αυτό το λόγο υποβάλαμε και απόρριψη, ε, τοπολογία περί αλλά θέλουμε να είμαστε και επικοδομητικοί και υποβάλαμε πολλές άλλες τροπολογίες για να δείξουμε το πώς βλέπουμε εμείς τα πράγματα. Πώς μπορεί να βελτιωθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Καταρχάς, θα θέλαμε να διατηρηθεί το σύστημα διοίκησης. Χρηματοδοτείται από κάτι μέλη το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Άρα διακυβερνητική ε, διοίκηση πρέπει να παραμείνει. Αυτό είναι και το λογικότερο. Δεύτερον, ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα δεν θα πρέπει να είναι μόνο ένα ταμείο διάσωση, αλλά να εστιάζεται επιβελτιώσεω σταθερότητα τη Ευρωζώνη. Αυτό χρειάζεται σήμερα η Ευρώπη και αυτό μπορεί να επιτευχθεί εάν γίνει υπεύθυνο το, το ESM για αυστηρότερη εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Χρειάζεται και καλύτερος έλεγχος των κρατών μελών και πρέπει να στιαθούμε εκ νέου στη βιωσιμότητα του χρέους και αυστηρού δημοσιονομικούς κανόνες. Ε, κλείνοντα. Είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε για βελτίωση του κειμένου. Αναφερθήκαμε στη σημασία του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και Δεθωτικών Μεταρρυθμίσεων και τη διατήρηση των προτεραιοτήτων των Εθνικών Κοινοβουλίων. Αυτά είναι βασικά θέματα για μας. Προσβλέπουμε σε συνεργασία με τους ηγητές από αυτού και με τους σκιώδεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ στους σκιώδεις ηγητές, στον σκιώδη του Άλντε θα δώσω το λόγο, στο Βολφ Κλίντς, αλλά δεν τον βλέπω. Άρα, σαν σκιώδης για την αρεσιμότητα, είχαμε επιμείνει αυτός ο μηχανισμός να έχει αναγκαία μέσα όταν αντιμετωπίσει καταστάσεις κρίσεων. Μηχανισμούς ε, οι οποίοι δεν ε, εφαρμόστηκαν όταν θεσπίστηκε το νόμισμα και όταν κυκλοφόρησε. Η ρεσιμότητα θα πρέπει λοιπόν να γίνεται περισσότερο εκ των υστέρων και όχι εκ των προτέρων. Όταν συμβαίνει κάποιο πρόβλημα, κάποια καταστροφή και πρέπει να βοηθηθεί μια χώρα που αντιμετωπίζει δυσκολίε, εν τί αυτή η περιπτώση τότε ξεκινά μια διαδικασία εφαρμογής διαθωτικών μεταρρυθμίσεων που συνοδεύουν τα υπόλοιπα μέτρα και πρέπει να υπάρξει και σύγκληση των νομοθεσιών σε τομείς φορολογικούς και κοινωνικούς για τα εθνικά κοινοβούλια και το ρόλο αυτών. Επιμένουμε ότι αν εγκαταφυθεί το ε, κεφάλαιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας δεν θα δώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο Ευρωπαϊκός Προπολογισμό τα χρήματα, αλλά οι προπολογισμοί εθνικοί ε, συνεπώς Πρέπει να υπάρξει συσχετισμός άμεσος μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων με τη διοίκηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Όσον αφορά την ονομασία, ε, πιστεύουμε ότι σωστό θα ήταν να διατηρηθεί μηχανισμός ευρωπαϊκός σταθερότητας, Δημοσιονομική σταθερότητας. Αυτό τον ορισμό και την ονομασία γνωρίζουν οι χρηματοπιστωτικές αγορές, άρα είναι άχρηστο να διατέξουμε τον κίνδυνο διατάραξης των αγορών αλλάζοντας το όνομα. Τέλος, όσον αφορά τον Υπουργό Οικονομικών, σημαντικό είναι να διαχωριστούν τα καθήκοντα του υπευθύνου του Eurogroup από αυτόν και αυτός υπεύθυνος να είναι υπουργό Οικονομικών και αυτός και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά να μην είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκονισμού Μηχανισμού Δημοσιονομικής Σταθερότητας. Είναι δύο καθήκοντα που πρέπει να είναι ξεχωριστά. Τούτων λεχθέντων. Δίνω το λόγο στον εκπρόσωπο των Πρασίνων, στον Σβέν Γκίγκολτ. Καλημέρα, Πρόεδρε. Καλημέρα. Πολύ σύντομα, υπήρξαν καρποφόρες συζητήσεις μεταξύ σκιωδών εισηγητών. Μόνο κάτι να τονίσω θέλω. Ποιες είναι οι βασικές μας προτεραιότητες. Άκουσα αυτά που είπε ο εισηγητής, ότι υπάρχει κοινή γραμμή, κοινή κατεύθυνση. Σε αυτή τη φάση των διαπραγματεύσεων το Κοινοβούλιο πρέπει να επικεντρωθεί κυρίως επί των δημοκρατικών και νομικών υποδομών και του σχήματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Αυτό είναι πολύ πιο αποδοτικό από το να επαναλαμβάνουμε τη συζήτηση που αφορά αλληλεγγύη, το πόσο στέρεος είναι ο μηχανισμός, αυτά εξυπακούονται για ένα τέτοιο ταμείο. Κατά το παρελθόν είχαμε πολλές διαφωνίες πάνω σε αυτά. Μπορεί να επαναληφθούν και εδώ. Αυτό δεν πρέπει να καταστρέψει τη δυνατότητα του Κοινοβουλίου να τοποθετείται σαφώς όσον αφορά την ευρωπαϊκή διάσταση των αποφάσεων. Το ESM από τη στιγμή που χρηματοδοτείται βασικά από τα κράτη-μέλη, από τον προπολογισμό των κρατών μελών, θα παραμείνει όσον αφορά τις βασικές αποφάσεις υπό την αιγίδα των εθνικών κυβερνήσεων και ελπίζουμε και υπό την αιγίδα των εθνικών κοινοβουλίων. Αυτό δεν πρέπει όμως να μας σταματήσει από το να απαιτούμε ξεκάθαρα δικαιώματα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να έχουμε λόγο όσον αφορά τα τεκτενόμενα. Γι' αυτό προτείναμε να έχουμε περισσότερα δικαιώματα όσον αφορά την επιλογή του διευθυντού, να ελέγχουμε το κατάλογο των υποψηφίων και με τα χαράς είδα ότι το ΕΛΚ υπέβαλε σχετικές παρόμοιες τροπολογίες. Θα θέλαμε επίσης το Κοινοβούλιο να την χάνει πλήρου απαλλαγή και να μπορεί τελικά να συμμετέχει στο ESM μέσω σχέσεω μεταξύ του ευρωπαϊκού προπολογισμού και του ESM. Τι ο τρόπος μπορούμε να ασκούμε δημοσιονομικό έλεγχο και τα συναφή δικαιώματα και αυτό είναι νομικό εφικτό άνευ αλλαγή του χαρακτήρα του όλου μηχανισμού που είναι κυβερνητικό. Πρέπει να έχουμε επίσης και ένα άλλο δικαίωμα. Σαν μέλη του Κοινοβουλίου και ατομικά θα μπορούμε να υποβάλουμε γραπτές ερωτήσεις. Ένα δικαίωμα που έχουμε όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή με τις εθνικές εποπτικές αρχές. Πρέπει να μπορούμε να αλλάξουμε και την δομή λήψεως αποφάσεων, ούτω ώστε όσον αφορά το προβλεπόμενο δίκτυο ασφαλείας, όσον αφορά το Ταμείο Διάσωσης Τραπεζών, οι αποφάσεις να λαμβάνονται γρήγορα, ούτω ώστε η κοινοβουλευτική έγκριση της πίστοσης στα κράτη-μέλη να μπορεί να ακολουθεί μια διαδικασία εκ των προτέρων, ούτως ώστε όταν μια ανάγκη παρουσιαστεί και είναι κατεπίγουση ανάγκη αποφάσεως, να μην υπάρχει πρόβλημα λόγω των υψηλών ορίων που προβλέπονται στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Είναι αξιόπιστο ένα δίκτυο ασφαλείας εάν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι πραγματικά σε περίπτωση κρίσης. Διαφορετικά δεν είναι αξιόπιστο μέτρο ασφαλείας και δεν μπορεί με αποτελεσματικό τρόπο να βοηθήσει τη σταθεροποίηση της τράπεζας και να βοηθήσει ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση. Τέλος πιστεύουμε ότι το Κοινοβούλιο στα πλαίσια της διαδικασίας απαλλαγής θα πρέπει να έχει πλήρη πρόσβαση στους ελέγχους όχι απλώς να εξετάζει τις εκθέσεις των ελεγκτικών φορέων, αλλά να έχουμε συγκρίσιμα δικαιώματα ελεγκτικά, όπως έχουμε με άλλα στοιχεία του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να μπορούμε να συμμορφωθούμε με το άρθρο 310 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, που προβλέπει μια ενιαίο χαρακτήρα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και όχι κατακαιρματισμό αυτού. Αυτά είναι θέματα που κανονικά πρέπει να τα εξετάζει και να εκφράζει σύμφωνη γνώμη το Ευρωκοινοβούλιο. Παρόλο που θα συνεχιστούν διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά την οικονομική πολιτική στα διάφορα κάτι μέλη. Στα πλαίσια συμβιβασμού ελπίζω να μπορέσουμε να ενισχύσουμε σημαντικά τα δικαιώματα του Ευρωκοινοβουλίου ε, προς την περιγραφή σα ε, κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ τους κοιόδης ηγητές για τη συνεργασία τους και ευχαριστώ και τους εισηγητές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ με τον κύριο Γίγκολτ. Η ομάδα της ΓΚΟΕ. Δεν βλέπω τον σκιώδη ηγητή της ΓΚΟΕ. Το EFTD. Ούτε από το ENF. Βλέπω κανέναν. Κύριε Μάνκα, μας είπατε ότι μας ενημέρωσαν ότι υπάρχει αδερμηνία από τα σλοβακικά. Αν και τα αρχικά σας λόγια, η αρχική σας εισήγηση ήταν πάρα πολύ σαφή. μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τη γλώσσα σας τώρα για να αναπτύξετε περαιτέρω το θέμα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, λοιπόν, κοιτάξτε, εκφράστηκαν κάποιες απόψεις. Ευχαριστώ πολύ για την ατμόσφαιρα που επικράτησε στις συζητήσεις. Πρέπει να πω πραγματικά ότι θέλουμε μαζί να λύσουμε τα προβλήματα που εντοπίστηκαν. Θα ευχαριστήσω ε, τους συναδέλφους για αυτά που άκουσα σήμερα. Τα περισσότερα κράτη-μέλη υποστηρίζουν μία ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αξιολογηθεί. Μετά μαζί μπορούμε να αποφασίσουμε και ποιο ε, ρόλο θα αναθέσουμε στο φορέα αυτό και τι ονομασία θα του δώσουμε. Και για τους ελέγχους και για την εποπτεία τι αρμοδιότητες θα δώσουμε για όλο το πρόγραμμα σταθερότητας. Ήδη σήμερα το ESM έχει αποφασιστεί και είναι ένας φορέας ε, σημαντικός για τις χρηματοπιστωτικές αγορές και έχει ένα κεφάλαιο στη διάθεσή του επαρκές. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή δεν ζητούμε άλλους πόρους, περισσότερους πόρους για το ESM. Προφανώς θα πρέπει να συμφωνήσουμε ε, επί του ονόματος του φορέα. Πώς θα μετονομαστεί το ESM. Δεν θα αλλάξουν όμως οι αρμοδιότητες συναρτήσει του ονόματος. Συμφωνώ με τους σκιώδεις ηγητές που είπαν ότι χρειάζεται μια εποπτεία από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από πλευράς Εθνικών Κοινοβουλίων. Πρέπει να καταλάβουμε μαζί, όλοι μαζί, ποια θα είναι η θέση αυτού του Ταμείου και θα πρέπει να συμφωνήσουμε επί του γεγονότος ότι το ταμείο αυτό θα είναι εκτός του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και δεν θα υπάρχουν έλεγχοι από το Ευρωκοινοβούλιο. Στο μέλλον όμως πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ίσως να, στο μέλλον υπάρξει και έλεγχος από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Αυτή την κατεύθυνση γενικώ επιθυμούμε. Όσον αφορά τα εθνικά κοινοβούλια, αναπτύσσεται η σημασία του ρόλου του όλο και περισσότερο έχουν όλο και πιο σημαντικό ρόλο τα εθνικά κοινοβούλια, διότι θα πρέπει να εγκρίνουν και το ρόλο αυτού του Ταμείου. Στο μέλλον, ίσως να μην έχουν πλέον αυτό το ρόλο, θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να ε, παγιώσουμε το ρόλο τους. Θα πρέπει να υπάρξει υποστήριξη για αυτό το μηχανισμό Εν πάση περιπτώσει ε, πρέπει να δούμε πώς θα ενημερώνονται τα εθνικά κοινοβούλια ούτως ώστε να μπορούν να έρχονται σε επαφή με τους διαχειριστές του Ταμείου να μπορούν να ασκούν ένα είδος εποπτείας στα κράτη-μέλη, τα εθνικά κοινοβούλια. Όσον αφορά ε, τους ε, συμμετρικούς και ασύμμετρους κλειδονισμούς, τα σοκ αυτά θα πρέπει να φροντίσουμε αυτό το ταμείο να βοηθάει την αντιμετώπιση των κλειδονισμών αυτών. Υπάρχουν και ασύμετροι κλειδονισμοί. Τι συμβαίνει όταν αντιμετωπίζει μια χώρα δυσκολίες. Αυτό είναι και ο ρόλος του Ταμείου, να λύνει τα διάφορα προβλήματα όπως αυτά ε, αναφύονται. Όταν δημιουργήθηκε όμως αυτό ο μηχανισμό, ε, αυτοί οι συμμετρικοί κλειδονισμοί οδήγησαν στο ότι πέντε κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν δυσκολίες. Η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Κύπρος, Ισπανία, Πορτογαλία. Και έτσι είδαμε και επανειλημμένα προβλήματα, αλυσιδωτά προβλήματα να εμφανίζονται. Πρέπει το Ταμείο να μπορεί να αντιμετωπίζει και συμμετρικούς κλειδονισμούς και ασύμμετρους. Αυτό το Ταμείο θα πρέπει να επιλύει σχεδόν εκ των υστέρων. Να αντιμετωπίζει περισσότερο τις συνέπειες. Να λειτουργεί περισσότερο εκ των υστέρων παρά εκ των προτέρων. Θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όμως όλες οι καταστάσεις και εκ των προτέρων εμφανιζόμενες και εκ των υστέρων. Καμιά φορά χρειάζεται να προλαμβάνουμε τις καταστροφές όταν οι αναλύσεις δείχνουν ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί κάποια κρίση. Συνεπώς θα, θα πρέπει οι χώρες να μπορούν να, έχουν, να δίνουν πόρους στο Ταμείο για να μπορούν να αντιμετωπίζονται αυτές οι αναταραχές, αυτοί οι κλειδονισμοί, αυτά τα σοκ. Αυτός ο μηχανισμός θα πρέπει να ενισχύει τη σταθερότητα των μελών του Ταμείου σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την πρόσβαση των κρατών στην πίστοση και στα, στις χρηματοπιστωτικές αγορές στην περίπτωση επιδείνωσης λοιπόν των προβλημάτων. Και αυτό μπορεί να γίνει αν κάνουμε μια καλή εκ των προτέρων ανάλυση. Θέλω για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης εισηγητές και στην τελευταία συνεδρίαση σημειώσαμε πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο και επί σημείων όπου ίσως δεν πιστεύαμε ότι θα συμφωνήσουμε. Λοιπόν, πραγματικά για μένα σημαντικό να συνεχίσουμε πάνω σε αυτή τη κατεύθυνση. Έχω την πεποίθηση ότι θα τα καταφέρουμε και ελπίζω ότι θα βρούμε τελικά μια συνένεση ούτως ώστε να καταλήξουμε σε μια καρποφόρα και καλή συμφωνία. Ευχαριστώ κύριε Μάκα. Ε, έχουμε λοιπόν λίγα λεπτά τώρα για τη διαδικασία κάτω στη ΆΗ. Μπερέση έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στο θέμα αυτό ξέρουμε πολύ καλά ότι το Συμβούλιο είναι αρκετά μπλοκαρισμένο, δεν προχωράνε τα πράγματα γρήγορα. Είναι λοιπόν σημαντικό ακόμα περισσότερο το Κοινοβούλιο να δώσει ένα μήνυμα μέσω των ε, εισηγητών αυτών και των ε, εκθέσεων αυτών. Και έτσι να δώσουμε τροφή για σκέψη στο Συμβούλιο. και να εξασφαλίσουμε τουλάχιστον ότι σε δύο-τρία θέματα θα λεφθεί υπόψη η απόψη του Κοινοβουλίου. Να επανέλθω λοιπόν και να αναφέρω δύο-τρία πράγματα. Το θέμα του ονόματο. Δεν θέλω να το ξανανοίξω το θέμα αυτό, αλλά με ικανοποιεί το γεγονό ότι είναι υποσυζήτηση με κάποιου ε, τύπου που μα φαίνονται αρκετά χρήσιμου ε, σε ό,τι αφορά το Ταμείο Ευρωπαϊκή Σταθερότητας. Θεωρώ ότι υπάρχει κίνδυνος ε, σύγχυσης με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αλλά θεωρώ ότι θα μας επιτρέψει να αλλάξουμε και τη φύση της δομής, περνώντας ε, από το μηχανισμό σε ένα ταμείο, σε ό,τι αφορά την μεταξέλιξη αυτή που προτείνεται. Εφόσον υπάρχει το status θεωρώ ότι θα μας ικανοποιήσει. Αυτό που όμως τελικά ε, δίνει ε, πραγματικά εμπιστοσύνη στις αγορές είναι να υπάρχει ισχυρή ευρωζώνη, ισχυρό νόμισμα, ισχυρή Ευρώπη χωρίς να χρειάζεται να υπάρχουν ε, έκτακτες καταστάσεις που δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη της οικονομίας. Πέρα τούτου σε ό,τι αφορά τις προθυμίες, την προθυμία και τι διαθέσει των αγορών, πιστεύω ότι θα βρούμε ένα συμβιβασμό σε ό,τι αφορά και την αρχική πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο θέμα τώρα των σχέσεων και το σύνδεση του ταμείου αυτού, του μηχανισμού αυτού και των συμφωνιών που ενδεχομένως να υπάρχουν μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμφώνου Σταθερότητα. Θα ήθελα να σα επιστήσω την προσοχή στο εξή. Μία παράγραφο η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων με μεγάλη πλειοψηφία και θεωρώ ότι εδώ το Κοινοβούλιο ενδεχομένω να σημειώσει μια αντίφαση, γιατί από τη μία έχουμε το σύμφωνο σταθερότητα μέσα στην συνθήκη και στόχο ε, δεν είναι άμεσα εφικτό, ε, άρα είμαστε σε μια ενδιάμεση κατάσταση. Αν ε, λοιπόν νομοθετήσουμε υπερβολικά τον ε, ε, μηχανισμό σταθερότητα ω ανεξάρτητο μηχανισμό πέρα από τις συνθήκε, ως μνημόνιο κτλ. Θεωρώ ότι η αυτονομία του οργανισμού τελικά θα μας αποτρέψει από τον απότερο στόχο που είναι η σύγκληση. Παράγραφος 7 λοιπόν, όπου οι συνεισηγητές ε, συμπεριλαμβάνουν το στις συμβιβασμούς. Πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ESM στέλνει το μήνυμα ότι θα αυξηθεί η αυτονομία του τελευταίου. Όταν άποψη του Κοινοβουλίου είναι ότι όπως προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ενωμητάξη Τάξη και στις συνθήκες. Τελευταίο σημείο, και αυτό πιστεύω ότι επίσης είναι πολύ ηχηρό μήνυμα που θα πρέπει να αποστείλει το Κοινοβουλίο, είναι η αρχή της πρόληψης, ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτή χωρίς πρώτερη αιρεσιμότητα. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά στοιχεία. Δεν θα ξαναξεκινήσω τη συζήτηση σε ό,τι αφορά την αλλαγή απόψεων που έχουν κάνει κάποιοι για την ε, αιρεσιμότητα, τους κανόνες, ε, τα περί μεταρρύθμισης, ερευνητικής μεταρρύθμισης. Θεωρώ ότι είναι σχεδόν ιδεολογική και φιλολογική αυτή τη συζήτηση. Δεν έχει κάποιο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι δεν θα βοηθήσουν την Οικονομική Ένωση όπως θα έπρεπε. Αν θέλουμε να δώσουμε στο ευρώ το ρόλο που την αναλογεί στην διεθνή σκηνή σε, όπως είπε και η Κεντρική Τράπεζα χθε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε την κυρία Περές. Άλλος κανείς. Ζητά το λόγο. Όχι. Να καλέσω λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παρουσιάσει και τις δικές της παρατηρήσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μας δίνετε το λόγο. Και θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω του συνεισηγητέ και του σκιώδει συζητητέ για τη δουλειά που κάνουν ω τώρα σε ό,τι αφορά αυτή την ε, διάμεση, το σχέδιο διάμεση έκθεση, σε ό,τι αφορά το ψήφισμά σα. Γενικά, προσυπογράφουμε το πνεύμα τη έκθεση και σημειώσαμε ότι η συζήτηση ήταν πολύ ζωηρή, όχι μόνο μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και στα, στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό πραγματικά μας χαροποιεί ιδιαίτερως. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας ωστόσο σε τρία στοιχεία τα οποία θεωρώ ότι προβάλλονται στην χρηματοδότησή σας. Καταρχάς, ε, εκτιμούμε την ε, υποστήριξή σας ε, στην έκκληση για την περαιτέρω ένταξη του ESM στο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. Κατά δεύτερον, όπως και το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή είναι υπέρ της ανακήρυξη τη ε, δημοκρατική ε, λογοδοσία. και τρίτον θεωρούμε ότι θα πρέπει να διευκρινιστούν με σωστό τρόπο οι ρόλοι του ESM είτε είναι η πρόταση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είτε είναι αυτή η ενδιάμεση φάση με να συνάδουν όλα αυτά με τις υπόλοιπες αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βασίζονται ακριβώς σε αυτό το νομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ. ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Πρόεδρε, θα μπορούσαμε να υποβάλουμε ένα ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόεδρος, βεβαίως, έχουμε 14 λεπτά στη διάθεσή μας ακόμα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχω μια απλή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από τις τροπολογίες των διάφορων πολιτικών ομάδων φαίνεται ότι πολλοί εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουν περισσότερα δικαιώματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τους ορισμούς, απαλλαγή κλπ. Γιατί όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προτείνει περισσότερα δικαιώματα ελέγχου για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πώς αυτό ταιριάζει με την Γενική Συμφωνία που έχουμε με την Επιτροπή Juncker κυρίως όταν πρόκειται για περισσότερη δημοκρατική εποπτεία από πλευρά του σώματο αυτού. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Να ακούμε την απάντηση της Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Γκίγκολτ. Αν προσέξετε τι ακριβώς προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, που ήδη είχαμε δημοσιεύσει το Δεκέμβριο του 2017, προβλέπεται ρόλος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, συμβουλευτικό για τον ορισμό του Γενικού Διευθυντή, αλλά Στο ESM, για παράδειγμα, επίσης υπάρχει η δυνατότητα να γίνονται κάποιες ακροάσεις και κλεισμένων των θυρών στη γραμμή που προτείνουν και άλλα σώματα τα οποία διασφαλίζουν την οικονομική σταθερότητα. Υπάρχει δηλαδή προσπάθεια να ενισχυθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα από εκεί και πέρα μπορούμε να δούμε αν αυτός ο ρόλος μπορεί να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο εφόσον το ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ωραία. Θα περιμένουμε τους ε, συνεισηγητές. Για να ακούσουμε ο κύριος Περέρα Σίλβα πρώτα απ' όλα τι έχει να πει. Αρχίζετε εσείς, έτσι, και ο κύριος Μακαμετά. Ωραία. Ευχαριστώ. Η ανταλλαγή απόψεων που είχαμε επιβεβαιώνει ότι υπάρχει περιθώριο για πολιτικό συμβιβασμό στον φάκελο αυτόν. Τώρα, επί της ουσίας. Να περάσουμε σε αυτό το πρότεινε ο συνάδελφος από το ΕΣΑΡ για την μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας προκειμένου αυτός να ελέγχει τη συμμόρφωση των χωρών μελών με τους δημοσιονομικούς κανόνες. Υπενθυμίζω αυτό που είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις τώρα, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην υπάρχουν επικαλύψεις στις αρμοδιότητες διαφορετικών οργάνων μεταξύ τους. Η οικονομική η εποπτή αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όταν έχουμε να κάνουμε με τα σχέδια προϋπολογισμού παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Eurogroup, μετά το Συμβούλιο. Δεν νομίζω ότι θα είχαμε να κερδίσουμε αν προσθέταμε άλλη μία φωνή στη διαδικασία αυτή. Εξάλλου υπάρχει ήδη ένα πρωτόκολλο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ESM για την οργάνωση της συμμετοχής στις διαδικασίες. Να αποφύγουμε πάντως επικαλύψεις μεταξύ των αρμοδιοτήτων του νέου φορέα και των ήδη υπαρχόντων οργάνων. Το θέμα δεν είναι η ξάντε αιρεσιμότητα, η εποπτεία και συμμόρφωση με τους σημερινούς δημοσιονομικούς κανόνες είναι ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ελέγξει. Βέβαια δημιουργούνται κρίσεις όταν υπάρχει ανάγκη για οικονομική αρρωγή τότε έχουμε να κάνουμε πολύ περισσότερο με την ex post αιρεσιμότητα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε, Πέντρο Σίλβα Περέιρα. Βλαντιμίρ Μάνκα τώρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Και το ελεκτικό συνέδριο επιβεβαιώνει ότι πρέπει να εφαρμοστεί διακυβερνητική λύση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ξέρουμε ότι αυτός ο μηχανισμός δεν χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Πρέπει να δούμε πώς θα γίνονται οι έλεγχοι του φορέα αυτού. Μπορούμε να θεσπίσουμε ίσως ένα ad hoc φορέα για να κάνει τους ελέγχους και αυτό για να σεβαστούμε το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μάνκα. Πρέπει να ακολουθούνται οι απλούστερες δυνατές ε, διαδικασίες και ο ρόλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, του Eurogroup και των διαχειριστών αυτού του μέσου να είναι σαφώ καθορισμένη, να μην υπάρχουν αλληλεπικαλύψει. Υπενθυμίστηκε σήμερα το πρωί, όσον αφορά τη χρηματοδότηση, πιστεύω ότι εθνικά κοινοβούλια πρέπει άμεσα να συμμετέχουν σε αυτόν. Πρέπει να υπάρχει να υπάρχουν εγγύησεις όσον αφορά δάνεια ή όταν πρέπει να υπάρχει αυστοποίηση κεφαλαίων η εθνική θα πρέπει οι εθνικοί προπολογισμοί να συνδράμουν και όχι ο ευρωπαϊκός. Δεν ξέρω αν τον έλεγχο το διεξάγει το ελεκτικό συνέδριο, ανεξάρτητη ελεκτική φορείς επιφορτισμένη που θα πιστοποιούν ε, τα οικονομικά που παρουσιάζονται, τους ε, λογαριασμούς και τους συλλογισμούς που παρουσιάζονται. Νομίζω ότι η κοινή συνεδρίαση της Μπότς και της ΕΚΟΝ μας επέτρεψε να κάνουμε διαπίστωση, άκρως ανθαρρυντική. Οι σκιώδεις εισηγητές θα συνεδριάσουν αύριο 30 Ιανουαρίου από τις 13 και 30 μέχρι 15 στην άθουσα ΑΣΠ 521. Και η επόμενη συνεδρίαση η κοινή θα γίνει 7 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες αλλά αυτή η συνεδρίαση θα πρέπει πρώτα να επιβεβαιωθεί τις επόμενες ημέρες θα λάβετε επιβεβαιώσει αλλά με μολύβι σημειώστε αυτή την πολύ πιθανή ημερομηνία. Στις 7 Φεβρουαρίου κοινή συνεδρίαση Bodge Econ. Άλλες ερωτήσεις υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Οπότε είναι πέραση συνεδρία σας.